No, no, no, se ve. Bueno, buenas tardes. Καλησπέρα σα. Καθίστε παρακαλώ. Καθίστε παρακαλώ. Γιατί θα ξεκινήσουμε την σημερινή μας συνεδρίαση. Σα καλωσορίζω όλους. Παρακαλώ ησυχία, λέει η Πρόεδρος. Παρακαλώ ησυχία. Ομάδα ΕΛΚ, παρακαλώ. Λοιπόν, καταρχήν έχουμε την υιοθέτηση της μερίσιας διάταξη σημείο πρώτο στην μερίσια, και πρέπει να σας ενημερώσω ότι έχουμε δύο αλλαγές. Η πρώτη αφορά το 8ο σημείο, την συμφωνία με το Μαρόκο, που μετά από έτοιμο του κυρίου Χάμλουντ που δεν είχε αρκετό χρόνο να διαβάσει την έκδοση στα αγγλικά η οποία στάλθηκε πριν από λίγε μέρες ζήτησε λοιπόν ο κύριος Χάγκλουντ να αναβάλουμε αυτό το σημείο που τον αφορά στην ημερήσια διάταξη. Αν συμφωνείτε λοιπόν και εσείς, θα εξετάσουμε το σημείο αυτό αργότερα. Και το δεύτερο αφορά το σημείο 10 της συνεδρίας των συντονιστών. Μετά από αίτημα ενός συντονιστή από την ομάδα των φιλελευθέρων, που σήμερα αποσιάζει επειδή συνοδεύει τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου στην Ιρλανδία. Ζήτησε λοιπόν να γίνει αύριο το απόγευμα η συνάντηση των συντονιστών μετά από την παρουσίαση από την κυρία Δαμανάκη του πακέτου μεταρρυθμίσεων. Μετά λοιπόν από την παρουσίαση της κυρίας Δαμανάκη στις 4.30 θα έχουμε τη συνεδρία των συντονιστών. Αυτά είχα να σας πω. Αν δεν έχετε παρατηρήσει σας προτείνω να υιοθετήσουμε την ημερήσια διάταξη όπως τροποποιήθηκε. και στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου θα δείτε τα στοιχεία που αφορούν τη συνεδρίασή μας. Έχουμε μετά το σημείο 2 της ημερήσία. τα πρακτικά, έγκριση των πρακτικών 15 και 16 6 Ιουνίου 2011. Αν δεν έχετε αντιρρήσει, εγκρίνουμε και τα πρακτικά. Τρίτον, έχουμε τι ανακοινώσει του Προέδρου στην ημερήσια διάταξη. Θα ήθελα να σα ενημερώσω ότι η συνεδρίαση της 31ης Αυγούστου που προβλέπεται για όλη την ημέρα θα γίνει τελικά μόνο το πρωί και περνάμε τώρα στις ψηφοφορίες. Καταρχήν έχουμε το σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης που αφορά... A ver, está... ψηφοφορία στο σημείο 4 παραλαμβάνει η Πρόεδρος, Σύμβαση για την διατήρηση και διαχείριση των λευτικών πόρων της ανοιχτής θάλασσας στο νότιο Ειρηνικό ωκεανό. Κυρία εσείς. Πρόεδρε, συγγνώμη, αλλά η κάρτα μου για την ψηφοφορία είναι στην άλλη επιτροπή που ήμουν πριν και μου τη φέρνουν τώρα. Τι να κάνω. Τίποτα. Μην κάνετε τίποτα. Εγώ θα ανακοινώσω τα αποτελέσματα, αλλά κάποτε θα πρέπει να τεθεί τέλος στην κατάσταση αυτή, επειδή το να ανακατεύουμε τις ψηφοφορίες δεν είναι κάτι βολικό. Η κυρία Ροντούς και ο κύριος Καντέκ θα πρέπει να σηκώσουν το χέρι και οι υπόλοιποι, αν συμφωνείτε, θα προχωρήσουμε έτσι. Α και δική σας δεν δουλεύει, αν θέλετε τότε να ψηφίσουμε όλοι με ανάταση, χειρός, γιατί δεν γίνεται να έχω τα μάτια μου 14. Τι θα κάνουμε λοιπόν. Για την πρώτη ψηφοφορία, επειδή είναι απλή, θα ψηφίσουμε διανάτες χειρός και μετά θα δούμε στη συνέχεια θα γίνει, αν περιπλεκούν ψηφοφορίες. Έκθεση φράγα. Δεν έχει τροπολογίες. Διαδικασία σύμφωνης νόμης. Οπότε θέτω σε ψηφορία την θέση της εισηγήτριας. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ε, ψήφι υπέρ, θα πρέπει να μετρήσουμε δυστυχώς. Ψήφι υπέρ. Και εμένα βάλτε έτσι. Κατά. αποχέ. Αποχές. Βρε για κοίτα, ομόφωνα. Για μια φορά συμφωνούμε όλοι εδώ στην Επιτροπή. Ομόφωνα ψηφίσαμε, μάλλον θα μπερδευτήκαμε θα ψηφίσαμε ομόφωνα. Ωραία, πάμε παρακάτω. Δεύτερη ψηφοφορία, Βαλέσα, για την πράσινη βίβλο που αφορά την έρευνα. Λοιπόν, ποιο δεν έχει κάρτα. εκτό από τους δύο, τρει μάλλον, τρει δεν έχουν ηλεκτρονική κάρτα, οι υπόλοιποι ψηφίζουμε ηλεκτρονική κάρτα. Καταρχήν, συμβαστική πρόταση 1. Ε, ψηφίζουμε. Πέρα της ψηφοφορίας. Ψήφισαν 18 συν 3. 21. 21 21 υπέρ, ομόφωνα. Εγκρίνεται η συμβαστική 1, οπότε καταπίπτουν η τροπολογία 2 και ψηφίζουμε την τροπολογία 3, η οποία αποτελεί προσθήκη. Ψηφίζουμε. Ναι, λέει η Πρόεδρος, ναι. Ναι, ναι, ψηφίζουμε. Πέρας της ψηφοφορίας 19 υπέρ και 2 κατά. Εγκρίνεται η τροπολογία 3. Η τροπολογία 1 καταπίπτει. Η 4 τώρα, τροπολογία 4. Ψηφίζουμε. Πέρα στις ψηφοφορίες, 21 υπέρ εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση 2. Ψηφίζουμε. Πέρας της ψηφοφορίας. Ομόφωνα και αυτή εγκρίνεται. Καταπίπτουν κατά συνέπεια η τροπολογία 5 και θέτουμε σε ψηφορία την τροπολογία 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Ομόφωνα και αυτή. Η 6 καταπίπτει η 7, καταπίπτει και η 8 και καταπίπτει και η εννέα. Ψηφίζουμε για την 10, τροπολογία 10. Άρχεται η ψηφορία. Πέρα στις ψηφοφορίες. Απορρίπτεται. Θέτω σε ψηφοφορία την τροπολογία 11. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα στις ψηφοφορίες. Απορρίπτεται. Θέτω σε ψηφοφορία τη συμβαστική πρόταση 3. Ψηφίζουμε. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Κατά πίπτουν οι 12, οι 14 και οι 26. Θέτουμε σε ψηφοφορία την τροπολογία 13. Άρχεται η ψηφοφορία. 13 λέει πρόεδρος. 13. 13. 13. compromiso 3 sí se sometido. Ah, la enmienda oral, es que hay una enmienda oral. Α, ah, δεν είχα σημειώσει εδώ. Έχουμε μια προφορική τροπολογία. Ναι, ναι, ναι. Να την είχα δει, λέει πρόεδρος. Συγγνώμη, συγγνώμη. Είχαμε μια τροπολογία προφορική που δεν την είχα στο, στο δικό μου κατάλογο ψηφορίας, δικό μου λάθος. Λέει πρόεδρος, συγγνώμη. Αλλά πρέπει να επανέλθουμε στην ε, προφορική Συμβαστική πρόταση 3, είναι μια προσθήκη. Ψηφίζουμε λοιπόν για την προφορική ε, τροπολογία 3, όπως ακριβώς αυτή έχει στο κείμενο. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται ομόφωνα. Καταπίπτουν λοιπόν οι 12, οι 14, οι 26, οι 24. Και θέτω σε ψηφορία τώρα την τροπολογία 13. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Θέτω σε ψηφοφορία τώρα την τροπολογία 15. Ψηφίζουμε. Πέρας της ψηφοφορίας. Έχουμε ένα του ΕΛΚ παραπάνω. Ένα του ΕΛΚ παραπάνω έχουμε. Και αυτό δεν έχει σχέση με τις ηλεκτρονικές κάρτες. να μην ψηφίσει ο κ. Τσουκαλά που είναι αναπληρωτή. Αναπληρωματικό μάλλον. Αλλά τι γίνεται με τον κ. Τσουκαλά. Τέλο πάντων, ψηφίζουμε θα, θα ψηφίσουμε ε, σε, στο όνομά σα μια συγκεκριμένη. Λοιπόν, ξεκινάμε για τη 15. 15, για τη 15. Τροπολογία 15. Πέρα τη ψηφοφορίας εγκρίνεται ομόφωνα. Συμβαστική πρόταση 4. Ψηφίζουμε. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται ομόφωνα. Καταπίπτουν η 16, η 19 και θέτω σε ψηφοφορία την 17 του κυρίου Τσουκαλά. Ψηφίζουμε. Πέρας της ψηφοφορίας Απορρίπτεται. Θέτω σε ψηφοφορία την τροπολογία 20. Ψηφίζουμε. Πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 13 εναντίον 8. Στη συνέχεια έχουμε μία προφορική τροπολογία υπαριθμών 1 του εισηγητή στην παράγραφο 4 να περιληφθεί η λέξη sufficient επαρκή. Αν υπάρχει προφορική τροπολογία ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε πέρα της ψηφοφορίας εγκρίνεται ομόφωνα. Θέτω στη ψηφοφορία την τροπολογία του 21. Ψηφίζουμε. Πέρα της ψηφοφορίας Απορρίπτεται. 18. Θέτω σε ψηφοφορία την τροπολογία 22. Ψηφίζουμε. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται ομόφωνα. 23 Φεραίρα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Πέρασε έτσι. Τελειώσαμε. Και αυτή εγκρίνεται ομόφωνα. Για την 25 ψηφίζουμε. Περάς. Απορρίπτεται. 27. Τροπολογία. Ψηφίζουμε. Περάς. Απορρίπτεται. Τροπολογία 28 ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 29. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 12.8. Τροπολογία 30. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 31. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 32. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 33. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 34. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 35. Τροπολογία. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 36. Χωριστά. Πρώτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Και το δεύτερο τμήμα με μια προφορική τροπολογία που διαγράφουμε το Mediterranean Black Sea Baltic. Baltic. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Περνάμε τότε στην τελική ψηφοφορία της νομοδότησης όπως τροποποιήθηκε. Ψηφίζουμε. Πέρας. Ομόφωνα 21 ψήφοι. Ομόφωνα. Συγχαρητήρια κύριε Βαλέσα. Και στερήσαμε και από το σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης. Πάμε τώρα στο σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης. Καταπολέμηση της παράνομης αλληλείας σε παγκόσμιο επίπεδο ρόλος της ΕΕ. Η κυρία Λοβίν είναι συγγήτρια θέμα που έχουμε συζητήσει επανελειμμένως. Σήμερα έχουμε προβλέψει μία συζήτηση για τις ε, τροπολογίες που έχουν κατατεθεί, οι οποίες είναι αρκετέ 122 τροπολογίες και θα δώσω το λόγο αρχικά στην κυρία Λόβιν για να ξεκινήσει την εισήγησή της και μετά θα δώσω το λόγο στους υποπούς βουλευτές. Κύριε Λόβιν, έχετε το λόγο. Ε, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας όλους τους σκιώδεις εισηγητές, όλους τους συναδέλφους που υπέβαλαν σε αυτές τροπολογίες, 122 από αυτές, και νομίζω αρκετά εντυπωσιακό αριθμό δείχνει πω η προσπάθεια καταβάλλεται στην Επιτροπή πάνω στο θέμα αυτό. Είναι πολύ σημαντικό θέμα που ήδη έχουμε συζητήσει. Εξαρτόμαστε πολύ βλέπετε από τις αγωγές και ο Ευρωπαϊκό Αλληλευτικό Στόλο δρά διεθνή ύδατα και έχουμε υποχρεώσει να δράσουμε. Έχουμε ευθύνη στον κόσμο. Έχω κάποια σχόλια επί κάποιων τροπολογιών που τις θεωρώ πολύ σημαντικές. Οι 32 και 33 πιστεύω ότι δεν είναι καλές Αναφέρεται εδώ η διαγραφή κάποιων λέξεων. Και λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να διστάσει από το να εντοπίζει και να υποστηρίζει τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όποτε αυτό θεωρείται ενδείκνητο όταν διακυβεύεται η εξοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαγραφή αυτών των λέξεων που προανέφερα θα είναι ατυχέστατο γεγονός για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα, όπως αναφέρει και η τροπολογία, διακυβεύεται η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν ζητάμε άλλα κράτη-μέλη και άλλοι φορεί να κάνουν πράγματα για να καταπολεμήσουν την παράνομη αλία θα πρέπει να κάνουμε και εμείς με τους δικούς μας υπηκόους και να είμαστε πολύ αυστηροί ρυθμίζοντας τα του οίκου μας. Υπάρχει κάτι, αυτό είναι προφανέστατο. Κάτι άλλο, όταν συζητήσαμε με τους εκπροσώπους των ΙΠΑ και της Ιαπωνίας εδώ, ε, είχα τη δυνατότητα να πιω καφέ μαζί τους, να γευματίσω μαζί τους, να κουβεντιάσω μαζί τους. Και τίθεται και το θέμα του ΠΟΕ. Αν έχουμε αυστηρότατο κανονισμό για την αλληλεία θα ζητάμε για κάθε ψάρι που σάγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση να συνοδεύεται από έγγραφο που δείχνει πώ αλλιεύθηκε και ότι είναι πραγματικά νόμιμο για να καταπολεμήσουμε την παράνομη αλία. Αν δεν είμαστε πολύ αυστηροί όσον αφορά τον εφοδιασμό τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω σε ψάρια, ίσω ε, να παραβούμε κανόνε του ΠΟΕ. Η Ρεμπέκα Λάντα από τη ΣΥΠΑ είπε ότι αυτό είναι το σημαντικότερο σημείο, σημαντικότερη παράγραφος της εκθέσεως. Πρέπει να είμαστε αξιόπιστοι και θα πρέπει να επιβάλλουμε κυρώσεις στα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Παρακαλώ να μείνει αυτή η διατύπωση στο κείμενο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τροπολογία 56. Έκανα μια μικρή διόρθωση του κειμένου μου εδώ λέμε ότι η καταπολέμηση της παρανόμου αλίας δεν είναι θέμα ελήψεως τεχνολογικών δυνατοτήτων ή πόρων αλλά κυρίως έλλειψης πολιτικής βουλήσεως για δράση. Και αυτό είναι σημαντικό, πρέπει να αναφερθεί. Κύριε Πετράου, είναι εδώ. Ίσως θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε λίγο την τροπολογία σας υπαριθμών 68. Εκεί αναφέρεται ότι η παράνομη αλία που γίνεται από τα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως είναι αποτέλεσμα κακής, κακά προσαρμοσμένης διαχείρισης κλπ. Ε, μπορείτε να διαβάσετε την τροπολογία μόνοι σας και ότι δεν, τα αλλιεύματα, τα ψάρια που αλλιεύονται δεν, αντιμετω, την πραγματική δυνατότητα που υπάρχει λόγω των, διαφόρων, των δυνατοτήτων που παρέχουν τα διάφορα είδη ψαριών. Κάθε αλλιεύς τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω θα πρέπει να σέβεται του κανόνε μα, εγώ αυτό πιστεύω. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα Ευρωπαίων αλλιέων που έχουν παραβεί συνειδητά κανόνες. Και έχουμε παράδειγμα με ένα σκάφος της Καναρίους νήσους που ψάρεψε παράνομα έξω από τη Σιέρα Λαώνα. Έχουμε περιπτώσεις στην Ιταλία. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Χρησιμοποιούν ε, δίχτυα παρασυρώμενα παρόλο που ε, απαγορεύονται δια και αυτέ οι δραστηριότητε ασκούνται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι ότι οι ψαράδε είναι αθώοι και ότι υπάρχουν πολλοί κανόνε και μπερδεύονται. Δεν ξέρω, μπορεί να το εξηγήσετε καλύτερα εσεί ίσω. Ε, τροπολογία 77. Μάλιστα. Τι θέλω να πω εδώ. Ίσως να θεωρηθεί υπερβολικό, ίσως αυτό να πιστεύετε, το ότι πιστεύω ότι εκεί που εκπροσωπούν συμβαλόμενα μέρη σε αντιπροσωπείες σε φορείς διαχείριση, περιφερειακής διαχείρισης αλίας θα πρέπει να δηλώνουν τα οικονομικά του συμφέροντα σε σχέση με τα λιεύματα ε, που διαπραγματεύονται. Γιατί αυτό είναι εύλογο. Διότι φορείς περιφερειακής οργάνωσης αλίας είναι οι μόνοι διεθνείς φορείς που ασχολούνται με ε, μεταναστευτικά ε, αποθέματα αλλιευτικά στο διεθνές επίπεδο. Και αυτά τα αλλιεύματα, αυτά τα είδη είναι η διευθυνσία της διεθνούς κοινότητος, δεν ανήκουν σε κανέναν και έχουμε την ευθύνη να διατηρήσουμε αυτά τα αλλιεύματα, αυτά τα είδη ε, και τώρα και για το μέλλον. οι αποφάσει που λαμβάνονται σε αυτό το τομέα δεν λαμβάνονται με αρκετή διαφάνεια. Άρα θα ήταν λογικό να ζητούμε ότι εκπρόσωποι χωρών που είναι συμβαλόμενα μέρη των συμφωνιών αυτών να είναι ε, αντικειμενικοί και να μην μεροληπτούν και να μην έχουν οικονομικά συμφέροντα όσον αφορά τα αλευτικά αποθέματα που συζητούνται και διαπραγματεύονται. Γι' αυτό υποβάλλουμε αυτή την τροπολογία και ελπίζω να μας υποστηρίξετε σε αυτό. Οι 93, οι 94 και οι 95 τροπολογίες αυτές φαίνεται ότι ίσως σκοπό τη διαγραφή της πρότασής μου. Δηλαδή να δημιουργηθεί νέος φορέας υπό την αιγίδα του ΟΗΕ που θα διεξαγάγει ανεξάρτητες αξιολογήσεις και για τις επιδόσεις των σκαφτό, σκαφών και για τις χώρες σημαίας. Ε, ίδια ιδέα είναι αυτή. Μιλάμε για την ιδιοκτησία της διεθνούς κοινότητας, για την καλή κατάσταση των ωκεανών του κόσμου. Ξέρουμε ότι εξαντλούνται τα αλλιεύματα, τα αλλιευτικά είδη σε σημαντικό βαθμό και χρειάζεται να έχουμε κοινό παγκόσμιο στόχο. Και η Επιτροπή Ελίας του ΦΑΟ δεν είναι ο φορέας εκείνος που μπορεί πράγματι να πάρει σκληρές αποφάσεις. Λοιπόν, και υποτίθεται ότι οι αρμόδιοι φορείς και τα σκάφη σημαία θα κάνουν, οι χώρες θα ελέγχουν τα σκάφη τους που φέρνουν τη σημαία τους όσον αφορά τη συμμόρφωση. Για το μέλλον, για να κινηθούμε σωστά, χρειαζόμαστε διεθνή μέσα για να γίνεται ανεξάρτητη εξολόγηση των επιδόσεων των διαφόρων οργανισμών που ασχολούνται με τη διαχείριση του διεθνούς πλούτου του αλλιευτικού. Γι' αυτό θα ήθελα να παραμείνει αυτή η διατύπωση στο κείμενο της εκθέσεως. Έχω και άλλα δύο σχόλια που αφορούν δύο άλλες ε, τροπολογίες. 96 είναι δική μου τροπολογία και αναφέρεται στο ίδιο. Δηλαδή, ότι υπάρχει προφανής έλλειψη διεθνού συνεργασίας όσον αφορά τη διαχείριση όλων των αρνητικών συνεπειών της ανθρώπινης δραστηριότητας πέραν της αλληλείας που οι δραστηριότητες αυτές επηρεάζουν το, το θαλάσσιο περιβάλλον. Βλέπουμε τα διάφορε ζυπαντικές ουσίε που φεύγουν από την Ευρώπη με τα ρεύματα αυτά στην Αρκτική γυρνάνε τον κόσμο, μολύνουν ε, ανθρώπους, αλλιεύματα στην άλλη άκρη του κόσμου. Βλέπουμε πλαστικά σκουπίδια που συγκεντρώνονται στο κέντρο του ειρηνικού. Αυξάνεται η οξύτη των υδάτων στους ωκεανούς ε, και απειλούνται τα κοράλια, τα οστρακόδερμα ε, αλλάζει το κλίμα και η δυνατότητα που έχει ο πλανήτης να απορροφά διοξείδιο του άνθρακο. Οι ωκεανοί του κόσμου είναι ο σημαντικότερος ρυθμιστής ε, του κλίματος. Είναι κρισίμου σημασία για την παραγωγή οξυγόνου, για τον άνθρακα, για την ανακύκλωση του νερού κλπ. Χρειαζόμαστε ολοκληρωμένη πολιτική σε παγκόσμιο επίπεδο για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Ταυτόχρονα. Γι' αυτό εγώ υπέβαλα την τροπολογία 96. Ήθελα να ακολουθήσω μια γενική σφαιρική προσέγγιση όσον αφορά το τι κάνουμε με το 72% της επιφάνειας του πλανήτη που είναι οι θάλασσες και οι ωκεανοί. Χρειάζεται κοινή προσέγγιση για να βοηθήσουμε τους πολίτες του κόσμου. Και τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους εκείνους που υπέβαλαν τροπολογίες που πρότεινα να έχουμε μια παγκόσμια βάση δεδομένων για το DNA. Είναι δυνατόν σήμερα. Θα είναι τεράστιο βήμα, σημαντικότατο για την ανιχνευσιμότητα των ψαριών στις παγκόσμιες αγορές. Αυτά είναι τα συγκεκριμένα μου σχόλια. Όπως σας είπα, είναι 122 οι τροπολογίες που υπευλήθησαν. Πολλά θέματα προς συζήτηση. Εγώ είμαι έτοιμη να ακούσω σχόλιά σας, παρατηρήσεις, ερωτήσεις σας και σας ευχαριστώ. Ε, Α, να πω κάτι. Θα προσπαθήσουμε να συντάξουμε συμβαστικές τροπολογίες. Να συναθρήσουμε τις τροπολογίες που αφορούν τον ίδιο τομέα και είναι αρκετές από αυτές που αναφέρονται στην ε, Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή, άλλε λένε ότι η παράνομη αλληλεία απειλεί την νόμιμη αλληλεία και του αλληλεί του τομέα, τους νόμους αλληλεί. Είναι ει βάρος αυτών και υπάρχουν και άλλες ε, τροπολογίες που μοιάζουν. Οπότε θα προσπαθήσουμε να προτείνουμε σχετικές συμβαστικές τροπολογίες. Ευχαριστώ. ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η καταπολέμηση της παράνομης και άνοχης αλίας είναι ένα δύσκολο πρόγραμμα και περιλαμβάνει σημαντικό έργο. Ε, συγχαίρω την Ιζαμπέλ για την ε, έκθεσή της και χαίρομαι ιδιαίτερος γιατί βλέπω το θέμα των εισαγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και των συνθήκων υπό τις οποίες γίνονται. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το συζητά στην έκθεσή της και αυτό είναι σημαντικό. Ελπίζω ότι θα μπορέσει να ε, συμπεριλάβει στην έκθεση το θέμα της ε, ανιχνευσιμότητας. Ξέρω ότι αυτό είναι σχεδόν αδύνατο να γίνει και υπάρχουν συνέπειες ε, αθέμη του ανταγωνισμού για τους ελλείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμη και αν, όπως είπε η Ιζαμπέλα, δεν είναι όλοι οι δικοί μας ελλείς οι πλέον αθώοι. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ δύσκολο να προσδιορίσουμε το μερίδιο της άναρχης αλίας στην αγορά μας και είναι σημαντικό να λάβουμε αυστηρά μέτρα όπως η απαγόρευση χορήγησης πιστοποιητικού εξαγωγής για χώρες των οποίων τα σκάφη γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι ασκούν τέτοια άναρχη και παράνομη αλία. Τέτοιου είδους μέτρα νομίζω ότι είναι σκόπιμο να τα προτείνουμε. Όπως έλεγε η Ιζαμπέλα Λεβίν ε, μόλις τώρα, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τους κανόνες ε, του ΠΟΕ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είχα πολλά να σας καθυστερήσω. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ κατέθεσα 11 τροπολογίες που αποβλέπουν στο να συμπληρώσουν και να διευκρινίσουν κάποιες πτυχές της έκθεσης που κατέθεσε η συγγήτρια τις οποίες στο γενικό προσανατολισμό συμμερίζομαι και ανταποκρίνοντας σε πέντε συγκεκριμένους στόχους. Πρώτος, είναι να προσπαθήσουμε να τοποθετήσουμε αυτό το πρόβλημα στην μέση διάταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν αφορά μόνο την αλληλευτική πολιτική αλλά και πολιτική εμπορική και ανάπτυξης και την εξωτερική πολιτική. Επίσης η εξέταση όλου του θέματος αυτού στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και αυτό ακριβώ το έκανα. Δεύτερον, Θέλουμε να διευκρινίζουμε πάντοτε όταν μιλάμε για την βιωσιμότητα. Η βιωσιμότητα περιλαμβάνει τρεις διαστάσεις. Η οικονομική, η περιβαλλοντική και η κοινωνική βεβαίως. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Οπότε τα θέματα αυτά αφορούν την κατάσταση των ωκεανών, βιοποικιλότητα, αλλά βεβαίως και τις ίδιες τις οικονομικές και εμπορικές πρακτικές που σχετίζονται με τον τομέα αυτό. Και το έκανα αυτό λοιπόν για να έχουμε μια πλήρη εικόνα. Τρίτο σημείο, τρίτος στόχος, η διαφάνεια. Αν θεωρούμε απαραίτητο να εντοπίσουμε τους ιδιοκτήτες των σκαφών και αυτούς που τα εκμεταλλεύονται και το θέματα των αδειοδοτήσεων. Για να αυξήσουμε διαφάνεια είναι σημαντικό λοιπόν να πούμε δύο λόγια σε αυτό το τομέα και έχουμε άλλη μια τέταρτη πτυχή η οποία αφορά στα θέματα που αφορούν τις χώρες, τις παράκτιες και τις χώρες ε, με τη σημαία. Και μια τελευταία πτυχή αφορά την τροπολογία 94 που μιλάει για την ανάγκη ύπαρξης μιας ε, πολυτομεακής προσέγγισης στα πλαίσια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και τα πόσο χρειαζόμαστε ιδιαίτερο οργανισμό εδώ ή όχι. Νομίζω ότι να υπάρχει πολυμερή προσέγγιση στα πλαίσια του ΟΗΕ είναι σωστό. Τώρα, κατά πόσο θα πρέπει να δημιουργηθεί να χρησιμοποιηθούν αντίθετα, οι υπάρχοντο οργανισμοί, νομίζω ότι αυτό ή να χρησιμοποιηθούν αντίθετα οι υπάρχοντες οργανισμοί, νομίζω ότι αυτό σαν συζήτηση είναι γενικότερο και ενδεχομένω θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα πρέπει να κάνουμε προσέγγιση αποσπασματική με την ύπαρξη πολλών ή πολλαπλών οργανισμών. Γι' αυτό ακριβώς ε, κατέθεσα την πρότασή μου που αποβλέπει ακριβώς σε αυτό, να αποτρέψουμε δηλαδή την υπερβολική αποσπασματοποίηση του πλαισίου των νομινόεθνων. Ευχαριστώ. Η κυρία Πατρόνια. Κυρία Πατρό, ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστούμε την Ιζαμπέλ και για τις εντατικές της προσπάθειες και γιατί μου ζήτησε να διευκρινίσω την τροπολογία μου. Η τροπολογία αυτή θεωρώ ότι είναι σημαντική. Θα προσπαθήσω να την εξηγήσω. Λέω ότι τμήμα της ελευθερικής προσπάθειας ε, που δεν είναι δηλωμένη ε, ε, Έχω ε, ε, στο νου μου ε, διάφορα αποθέματα. Όπως το προσφυγάκι, παραδείγματος χάρη. Και το τάκ για το προσφυγάκι δεν είναι επαρκές. Αυτό είχα κατά νου πίσω από αυτή την τροπολογία. Δηλαδή, αφενός μεν η μέθοδος διαχείρισης δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και οι αλληλείς δεν μπορούν να κατανοήσουν καθόλου τις αποφάσεις που λαμβάνονται στις Βρυξέλλες ε, μακριά από την πραγματικότητα. Γιατί οι αλληλείς βλέπουν ε, το πώς έχουν τα πράγματα επιτόπου. Υπάρχει λοιπόν ένα πρόβλημα επικοινωνίας το οποίο πρέπει να ξεπεράσουμε. Και αυτό το πρόβλημα επικοινωνίας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα διότι είναι εις βάρος της αλίας και επιδεινώνει την κατάσταση, ακριβώς αυτή την κατάσταση που θέλουμε να αποφύγουμε. Επίσης χρειάζεται να επανέλθει η αλληλευτική πολιτική πιο κοντά στις περιφέρειες για να είμαστε πιο κοντά στους πολίτες και να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα που τους πλήττουν να δούμε τον οικονομικό χαρακτήρα των προβλημάτων και να αναλάβουμε την κατάλληλη δράση. Είναι λοιπόν διτή η κατεύθυνση προς την οποία θέλω να κινηθούμε και αυτό θέλω να εκφράσω με την τροπολογία μου. Θα μπορούσαμε να αλλάξουμε κάπως τη διατύπωση της τροπολογίας μου για να μην υπάρχει καμία παρανόηση, αλλά αυτό είναι το μήνυμα το οποίο ήθελα να σας περάσω. Ευχαριστώ, κύριος Ντέβις. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Υπάρχει νομίζω μεγάλη υποστήριξη από την Επιτροπή για καταπολέμηση της παράνομης αλίας που βεβαίω ε, πλήττει τα αλληλεύματα και υπονομεύει τους νομιμούς αλληλευτές. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει το μήνυμα της Επιτροπής μας γνωρίζοντας ότι τα μέτρα που θα εφαρμόσουμε σχεδόν ε, σίγουρα θα υποστούν αποδυνάμωση και συμβασμούς πριν υιοθετηθούν οριστικά. Οι 70 και 100 τροπολογίες που αφορούν τα τρίτα μέρη νομίζω είναι θετικές και να αναφερθώ σε αυτό που λέει η Ιζαμπέλα για την τροπολογία 32 και 33. Δεν είμαι βέβαιος κατά πόσο έχουν θέση εδώ γιατί νομίζω εδώ εκθέτουμε τους, υποψη... τους υπεύθυνους συγγνώμη, και λέμε ποιοι ακριβώς είναι αυτοί που κάνουν τις παράνομες δραστηριότητε. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχουν κάποιοι οποίοι διπράττουν κάποιες παρανομίες θα πρέπει να πούμε ποιοι είναι αυτοί και να σταματήσει αυτό το φαινόμενο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ναι, να πω ότι είναι σημαντική αυτή η έκθεση. Γεννά πολλές προσδοκίες και αφορά πολλές δυνατότητες. Γι' αυτό ακριβώ έχουμε 122 τροπολογίες. Νομίζω ότι είναι μια από τις εκθέσεις που έχει τις μεγαλύτερες παρουσιάσεις και συζητήσεις λόγω της σημασία της. Υπάρχουν λοιπόν σημαντικά στοιχεία εδώ και θα πρέπει να ενισχυθούν. Καταρχήν θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει την θέση ηγετική που έχει για την καταπολέμηση αυτού του ενδημικού και δύσκολου προβλήματο, Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση τόσο όσον αφορά τα χωρικά υδατά της όσο και μέσω των εθνών συμφωνιών θα πρέπει να διασφαλίζει την αποτροπή τη παράνομη αλληλεία. Αυτό νομίζω είναι βασικό ως αρχή. Επίση έχουμε ένα σημαντικό στοιχείο συντονισμού μεταξύ των διαφόρων δομών και αγορών, κάτι το οποίο είναι επίση πολύ σημαντικό. Ή έχουμε επίση να κάνουμε και με το θέμα των συνόρων, θέμα πολύ δύσκολο να ρυθμίσουμε και το οποίο προκαλεί προβλήματα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαφάνεια για τη δημοσίευση των στοιχείων είναι θέμα σημαντικό και θα πρέπει να ενισχυθεί. Επίση, θα πρέπει να ενισχυθούν τα στοιχεία που αφορούν τι υποχρεώσει τόσο όσον αφορά τι δράσει αλλά και τι κυρώσει. Και βεβαίω, κυρίω το θέμα του ελέγχου τη ε, φορολογική απάτη, κατά το οποίο αυτή τη στιγμή αφορά ε, διάφορα και ποικιλόμορφα θέματα τη στιγμή που είναι προφανές ότι υπάρχουν θέματα φορολογικής απάτης και στην Ευρώπη αυτά τα θέματα, μάλλον αυτές τις πρακτικές προστατεύονται, οπότε θα πρέπει εδώ να λέμε ξεκάθαρα ότι αυτά θα πρέπει να υπάρχουν, να υφίστανται στον τομέα της αλληλείας. Οπότε καλές 122 τροπολογίες και νομίζω ότι είναι πολύ καλό αυτό που έκανε η εισηγήτρια να αποδεχτεί πολλές συμβαστικέ τροπολογίες. Μιλήσαμε συγκεκριμένα για τα προσφυγάκια θέμα που επανέρχεται. Εντάξει, υπάρχουν και άλλοι λιμένες και αυτό ακριβώς είναι σημαντικό να υπάρχει διαφάνεια και ύπαρξη δημοσιευμένων στοιχείων που να αποδεικνύει ακριβώς ότι υπάρχουν και άλλα λιμάνια που αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα. Αλλά να πω επίσης ότι και πριν από λίγες μέρες είχα μια συμφωνία μεταξύ Γενικής Διεύθυνσης Αλίας και Γενικής Διεύθυνσης θελωνίων στην Ισπανία για να προσπαθήσουν ακριβώς να αλλάξουν αυτό το πρόβλημα που ανακύπτει σε λιμένες οι οποίοι είναι πολύ μακριά από την Ευρώπη. Και αυτό ακριβώς αφορά τα όρια και τα σύνορα της ίδιας Ευρώπης και γι' αυτό ακριβώς θεωρώ το θέμα διαφάνειας είναι πολύ σημαντικό. Αν δεν υπάρχει κάποιο άλλο, η κυρία Λόβιν. Α, όχι. Η Κομισιό νομίζω, λυπάμαι πολύ που σας ξέχασα, δεν σα ξέχασα ακριβώ. Σας είχα και στην άκρη του ματιού, αλλά ξανά σα δώσω το λόγο. Έχετε πάντως το λόγο. Ε, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλω να υποστηρίξω την έκθεση τη κυρία Λαβίν. Θεωρούμε ότι 122 τροπολογίες καταδεικνύουν τον ενθουσιασμό και τη σημασία που έχει αυτή η έκθεση. Είμαστε υπέρ των μέτρων που ενισχύουν την καταπολέμηση της παρανόμου αλληλείας και σε διεθνές και σε εσωτερικό επίπεδο. Οι περισσότερες τροπολογίες ενισχύουν αυτή την ιδέα και νομίζω ότι κινούμεθα προς την κατεύθυνση που επανειλημμένα ανέφερε η κυρία Δαμανάκη. Δηλαδή ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει συνοχή μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής προσεγγίσεως. Συμμεριζόμαστε λοιπόν τις ιδέες των τροπολογιών όσον αφορά την ενίσχυση των προσπαθειών που καταβάλουν τα κράτη-μέλη και την ενίσχυση των διαφόρων φορέων διαχείριση τη αλληλεία. Προ αυτό το σκοπό είμαστε υπέρ μηδενική ανοχή όσον αφορά τι αγωγικέ προϊόντων που έχουν αληθεί παράνομα. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πολλοί το υπογράμμισαν από του προλαλήσαντε και ο ρόλο του κοινοτικού οργανισμού του αρμόδιου φορέα είναι πάρα πολύ σημαντικό Αύριο ίσως μπορούμε να το συζητήσουμε περαιτέρω με, το νέο, ε, με τον νέο διευθυντή το θέμα. Η συζήτηση είναι ανοιχτή. Πρέπει να συνεχιστεί. Είμαστε υπέρ κάθε μέτρου που θα μπορούσε να ενισχύσει την καταπολέμηση της, ε, αυτής της παρανόμου και αδήλωτης αλίας. Από την κυρία Θαμανάκη ζητήσαμε επανειλημμένως να δείξει περισσότερη πολιτική βούληση για την εφαρμογή του 2005. Έχω αμφιβολίες βεβαίως για την εφαρμογή του 2005 σε πολλές περιοχές όπως ο Ρηνικός, αλλά εφόσον η έλεγχη είναι ελλειπής, να πω και στο συγγνώμη ότι έχω αμφιβολίες για αυτά που λέει η Επίτροπος, γιατί βλέπω να λείπει η πολιτική βούληση σε αυτό το θέμα. Κύριε Λοβίν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους τους ε, συναδέλφους, σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας και για τις ε, εξηγήσεις σας. Νομίζω ότι θα έρθω σε επαφή με εκείνους από εσά που θέλετε να συμμετάσχετε στη διαμόρφωση συμβαστικών τροπολογιών και θα ψηφίσουμε μετά το καλοκαίρι. Οπότε δεν βιαζόμαστε. Άρα θα επανέλθουμε τον Αύγουστο, αρχές Σεπτεμβρίου στο θέμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Είχαμε προβλέψει την ψηφορία στην Επιτροπή στις 19 του Σεπτέμβρη. Θα έχουν επιτευχθεί απαραίτητοι συμβασμοί εκ μέρου τη κυρία Λεβά, νομίζω, μέχρι τότε και θα περάσουμε στην ψηφορία. Ωραία. Τελειώσαμε και με το σημείο 6 τη ημερήσια διάταξη. Η κυρία Ρέιμερ απουσιάζει για το σημείο 7. Οπότε, τι έγινε, θα τη τηλεφωνήσετε. Άντε, τηλεφωνήστε τη γιατί πέντε λεπτάκια θα περιμένουμε. Το 8 αναβλήθηκε, θα πρέπει να περιμένουμε λοιπόν την κυρία Ρέιμες 5 λεπτάκια διάλειμμα για να κάνετε βόλτα να βγείτε έξω στα πλαίσια της αναρχικής αυτής επιτροπής. Άντε, πέντε λεπτάκια διάλειμμα λέει η Πρόεδρος.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 Okay. Ήρθε η κυρία Ρέιμερς, μπορούμε να αρχίσουμε. Παρακαλώ καθίστε. Θα ξεκινήσουμε την συνεδρίασή μας και πάλι. Παρακαλώ. Κυρία Πατράου και η κυρία... Δεν λέει η Πρόεδρος. Είμαστε στο 7 θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο προπολογισμού 2012 όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο. Η συγγήτρια κυρία Ρέμερ, έχετε το σχέδιο γνωμοδότησης στου φακέλου σα και νομίζω έχετε λάβει και τα τελευταία στοιχεία από το Κορεπέρ που θα πρέπει να εθετηθούν από το Συμβούλιο. Έχουμε λοιπόν και εδώ τα διαθέσιμα τα στοιχεία του Κορεπέρ και θα δώσω το λόγο στην κυρία Ρέιμερς για να μας παρουσιάσει τη γνωμοδότησή της. Ευχαριστώ πολύ. Ε, καταρχήν ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά είχαμε στην Επιτροπή Γεωργίας ε, την ε, συνάντηση με τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων για την, ε, γεωργική για την αγροτική μεταρρύθμιση και δεν ήθελα να λείπω. Λοιπόν, για την γνωμοδότησή μου τώρα. Θα ήθελα να τονίσω τρία σημεία από το κείμενο της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Υπάρχει το κείμενό μου και υπάρχουν και τα πιλωτικά προγράμματα. Καταρχήν για τη δική μου γνωμοδότηση. Γνωρίζουμε ότι ε, πρέπει ε, αυτά που συζητάμε να τα συζητάμε στο πλαίσιο των μειωμένων πόρων γενικότερα. Και στον τομέα της γεωργίας ε, υπάρχουν σημεία κλειδιά για την οικονομία πολλών περιοχών και για ολόκληρη την Ευρώπη. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να φροντίσει τους πόρους της σε αυτό το τομέα και να διατηρήσει το επίπεδο των δαπανών σε τέτοιους τομείς ώστε να ενισχύσει την οικονομική δραστηριότητα. Έχουμε τις ε, περιοριστικές προτάσεις που έχουν υποβληθεί και με βάση ε, ε, τα στοιχεία που έχουμε θέλουμε να, να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί. Πιστεύω ότι θα πρέπει η Επιτροπή να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις όσον αφορά τις ε, πιστώσεις πληρωμών και αυτό μπορεί να μας το εξηγήσει ο εκπρόσωπος της Επιτροπής εδώ. Και στο σημείο 5 θέλουμε να μιλήσουμε για τους πόρους που δίδονται στον Οργανισμό για την Αλία με βάση αριθμητικά στοιχεία. Τώρα, όσον αφορά συγκεκριμένα, τα συγκεκριμένα σημεία, ε, Δεν μπορούμε πάντοτε να ζητάμε περισσότερα χρήματα, το ξέρουμε. Υπάρχουν όμως και εξαιρέσεις. Στο σημείο 11.01.04.03 Μιλάμε για στήριξη της διοίκησης των αλλιευτικών πόρων. Εδώ, ιδίω για την συλλογή δεδομένων και για τη βελτίωση των επιστημονικών αναλύσεων. Στον τομέα αυτό, η Επιτροπή έχει και εξωτερικές ε, υποχρεώσεις ε, και γι' αυτό πρέπει να παραμείνουμε σε αυτό το ποσό και να μην δεχθούμε μειώσεις. Το 11.02.03 και 04 ε, συμφωνούν η Επιτροπή και η Κορεπέρ, η Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων, και μετά περνάω στο 11.06 στο Ταμείο για την Αλία. Εδώ η Κορεπέρ προτείνει μείωση 8,3%. Μου κάνει εντύπωση, διότι εδώ πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενες πιστώσεις με τα κράτη-μέλη. Ε, και εδώ θα υποβάλει μια τροπολογία ώστε να παραμείνουν οι αρχικά, οι αρχικά προβλεπόμενοι πόροι. Το ίδιο ισχύει και για το 11.07. Εδώ ήδη είχαμε περικοπές το 2011 και θα πρέπει να αποκατασταθεί ο προϋπολογισμός στο αρχικό του επίπεδο. Στο κεφάλαιο 11.08 έχω ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η έλεγχη και η επιβολή της κοινή αλληλευτικής πολιτικής ε, είναι ένα σημαντικό θέμα και εδώ δεν πρέπει να κάνουμε οικονομίες. Θα πρέπει να αποκαταστήσουμε το αρχικά προτινόμενο ποσό τουλάχιστον αν δεν ζητήσουμε και περισσότερα. Και αυτό θα προσπαθήσω να επιτύχω με τις τροπολογίες μου. Περνάω τώρα στα πιλωτικά προγράμματα. Τα δύο πιλωτικά προγράμματα αξιολογήθηκαν θετικά από την Επιτροπή. Είναι μια προσπάθεια για περαιτέρω έρευνα για το θαλάσσιο χώρο. Σας παρακαλώ, αγαπητοί συνάδελφοι, να υποστηρίξετε ε, τις προτάσεις μου για τα πιλωτικά προγράμματα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ, λέει ο κύριος Βαλέσα. Κυρίες και κύριοι, συμφωνώ με τα όσα είπε η προλαλήσασα και την απεσιόδοξη προσέγγιση, αλλά μήπως έπρεπε να είμαστε πιο αισιόδοξοι στο τέλος. Συμφωνώ, σε αυτή τη φάση περνάμε σε παγκόσμιο επίπεδο μια οικονομική κρίση και είναι στιγμή για οικονομίες, αλλά οι συζητήσεις για τις οικονομίες δεν θα πρέπει να εδράζονται επί των τεκτενωμένων στι αγορέ. Θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε τι ευκαιρίες που μας δίνει η αγορά, το εμπόριο. Να δούμε πώς μπορούμε αυτά που κάνουν τον προπολογισμό να τα χρησιμοποιήσουμε για οικονομική ανάπτυξη. Να δούμε την ε, φωτεινή πλευρά των συζητήσεων για την οικονομία. Να δούμε τι καλό μπορούμε να δώσουμε στους πολίτες. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να μιλήσουμε για την χρηματοδότηση της αλίας. Στις 24 ώρες θα δούμε το νέο πακέτο για την κοινή αλληλευτική πολιτική. Προφανώς η μεταρρύθμιση θα είναι μεγάλη, ευρεία, θα χρειαστεί ε, πόρους, αρκετούς πόρους και δεν χρειάζεται να πείσω κανέναν από εσά ότι για να εφαρμοστεί αυτή η πολιτική χρειάζονται πόροι. Η αλληλευτική πολιτική περίμενε ε, επί και μεγάλο χρονικό διάστημα για την ευκαιρία αυτή θα δίδετο. εδίδετο. Και δεν θα πρέπει να μην εφαρμοστεί ένα τμήμα του πακέτου λόγω λήψεω πόρων. Υποστηρίζω αυτά που λέει η γνωμοδότηση για τις περικοπές, τις δαστικές περικοπές σε κάποιου τομείς ε, που γίνονται και χρειάζεται υποστήριξη ο τομέας που ήδη υποχρηματοδοτείται. Περικοπές στον τομέα Οι περικοπέ δεν θα μας επιτρέψουν να έχουμε ισορροπημένη ανάπτυξη αλληλεία στην Ευρώπη. Ούτε να προωθήσουμε την ισορροπημένη αλληλεία στον κόσμο. Ένα παράδειγμα εδώ είναι οι συμφωνίε που συνάπτουμε με τρίτε χώρε. Υπέχουμε κάποιε οικονομικέ υποχρεώσει εναντίον των εταίρων μα. Ερώτηση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν οι περικοπέ εγκριθούν σε αυτό το τομέα, εμεί πώ θα ανταποκριθούμε στι υποχρεώσει που έχουμε αναλάβει. Η κατάσταση αφορά τα κονδύλια για την αλία είναι η εξή. Περικοπέ, περικοπέ και ξανά μανά περικοπέ. Άρα δεν θα έχουμε τελικά χρήματα αρκετά για να καλύψουμε όλα όσα θέλουμε. Και κάτι που ανέφερε η συγγήτρια για τα πιλωτικά προγράμματα. Υπάρχει πιθανότητα να παρουσιαστούν, να υποβληθούν. Ποια είναι η άποψη του Συμβουλίου γι' αυτό. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την συγγήτρια. Θα ήθελα να καταθέσω δύο τροπολογίες που θα ήθελα να κάνουμε. Η υπηρεσία ελέγχου της Κομισιόν αφορά η πρώτη, όπως είπε η συγγήτρια, που θα ήθελε να επαναφέρει τις περικοπές για αυτή την υπηρεσία. Συμφωνούμε γι' αυτό. Και υπάρχει επίσης και ένα άλλο συγκεκριμένο αίτημα εδώ σε σχέση με τις δυνατότητες της Υπηρεσία ελέγχου για την υλοποίηση των συμβάσεών της όσον αφορά την εποπτεία στα διεθνή ύδατα στο ΕΚΑΤ και στον ΝΑΦΟ. Μιλάμε για την ενοικίαση σκαφών ελέγχου. Αυτό είχε περικοπεί από αυτό τον προπολογισμό. 4 εκατομμύρια ευρώ είχαμε στον προπολογισμό για το περσινό έτος που αποουσιάζει από το φετινό προπολογισμό. Η ιδέα λοιπόν είναι ότι η υπηρεσία αυτή θα πρέπει να ζητήσει οικονομική ενίσχυση από τις χώρες μέλη για να επιβλέψει ακριβώς την εφαρμογή των υποχρεώσεων των σκαφών αυτών. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει λόγω της κρίσης αμφιβολία κατά πόσο θα συμβάλλουν χωρίς μέλη στην υλοποίηση αυτή που αφορά τα σκάφη ελέγχου και νομίζω ότι γι' αυτό ακριβώ το λόγο θα πρέπει να χρηματοδοτούνται τα σκάφη αυτά από τον προπολογισμό της ε, κοινότητας. Νομίζω ότι αυτό είναι ουσιώδε όσον αφορά την δική μας ελευτική πολιτική, ώστε να συντονίσουμε τις προσπάθειές μας από τη στιγμή που τα σκάφια αυτά ελέγχου θα καθοδηγούνται και θα προερχόνται από την, Επιτροπή, από την υπηρεσία ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι ο έλεγχος και οι δικασίε ελέγχου και υποπτία είναι κάτι το οποίο μα βρίσκει σύμφωνο σε όλου. Να πω και δύο λόγια σχέση με τα πιλωτικά προγράμματα. Γνωρίζουμε όλοι ότι βρισκόμαστε στα μέσα της ανθεώρησης της κοινή ελευθερικής πολιτικής και εδώ έχουμε να κάνουμε και με τις εξωτερικές πτυχές της αληθικής πολιτικής. Ξέρουμε ότι η Κομισιόν θα προτείνει και είναι και αυτό διεθνής υποχρέωση ότι μπορούμε να αλλιεύουμε μόνο από τα πλεονάσματα των αλλιευμάτων. Επιστημονικώς αποδειγμένα πλεονάσματα. Όμως ε, δεν θα πρέπει να υπάρχει έλλειψη επιστημονικών στοιχείων για αυτά τα πλεονάσματα. Προτείνουμε λοιπόν 2 εκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση πλεοντικών προγραμμάτων που θα αφορούν ερευνητικά προγράμματα, επιστημονικά ερευνητικά προγράμματα στη Δυτική Αφρική και βεβαίως θα υπάρχουν και τα απαραίτητα σκάφη τα οποία θα κάνουν τις ε, έρευνες για είδη που δεν είναι ε, τόνοι. Και νομίζω αυτό είναι και το κύριο πρόβλημα εδώ. Θα ήθελα λοιπόν να αφιστήσω την προσοχή σας στο λόγο για τον οποίο έχουμε φτάσει στην τωρική κατάσταση. Έχουμε ένα νορυγικό σκάφος το οποίο κάθε τρία χρόνια περνάει από διάφορες περιοχές και οι αποτιμήσεις των αλλιευμάτων, των αποθεμάτων μάλλον, δεν είναι ιδιαίτερα αξιόπιστες. Αν θα πρέπει λοιπόν να έχουμε σωστές συμφωνίες, χρειαζόμαστε καλύτερα επιστημονικά στοιχεία και αυτό εδώ αποτελεί μια θαυμάσια ευκαιρία χρήσης των χρημάτων των φορολογουμένων για να έχουμε μια σωστή επιστημονική ενημέρωση για τα αποθέματα. Αυτά θα λοιπόν καθέσω αυτές τις τροπολογίες. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Κατέκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω καταρχήν να συγχαρώ την Πρίτα για τη γνωμοδότησή τη για το σχέδιο προπολογισμού για το 2012 και θέλω να πω ότι συμφωνώ με τα περισσότερα από τα σημεία τη γνωμοδότησή τη. Ε, χαίρομαι ε, για τον προπολογισμό που προτείνει για το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθηση των ε, Τιμών των Αγορών και συμφωνώ με την εισηγήτρια ότι είναι κρίμα να μειώνουμε τις πιστώσεις υποχρεώσεων και πληρωμών για θέματα ελέγχου όπως ε, ανέφερε και η Ιζαμπέλ. Υπάρχουν διαφορές σε θέματα ελέγχου σε επίπεδο διαφορετικών κρατών μελών ε, και αυτό δημιουργεί προβλήματα. Δεν πρέπει όμως να μειώσουμε τις δαπάνες. Ενδεχομένω πρέπει να βρούμε κάποιους άλλους πόρους. Όπως και η Μπρίτα, ε, συμφωνώ και εγώ για τον ε, προϋπολογισμό της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής και ακούσαμε και την έκθεση της Επιτροπής ε, για τα πιλωτικά προγράμματα. Ε, δεν ξέρω αν ε, κατά τύχη συζητήθηκαν αυτά τα θέματα και την περασμένη εβδομάδα και τώρα. Πάντως απορρίφθηκαν τα περισσότερα από τα άλλα προγράμματα, ενώ για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική υπάρχει υποστήριξη της Επιτροπής. Δεν θα πρέπει να μειωθεί λοιπόν ο προϋπολογισμός υπολείπων προγραμμάτων για να υποστηρίξουμε την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική και στο πολιτές πρόγραμμα προβλέπει ένα κοινό ταμείο η Επιτροπή για την περίοδο 2013-2020 και θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα ώστε αυτός ο προϋπολογισμός ε, να λαμβάνει πλήρως υπόψη την πολιτική αλίας. Αυτά για την έκθεση της κυρίας Ράιμερς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια για τη γνωμοδότησή της την υποστηρίζω και χαίρομαι που ε, εκφράστηκε κατά των περικοπών που έχουν προταθεί. Ε, βρίσκεται μια μεταρρύθμιση υπό επεξεργασία, υπάρχουν πολλά νέα στοιχεία ε, και η περικοπή 6,8% θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα λυπηρή. Και είναι κρίμα που περικοπές προτείνονται στα θέματα συλλογής δεδομένων που είναι γύρω στα 6,2% και όπως όλοι γνωρίζουμε υπάρχει μεγάλο έλλειμμα σε θέμα δεδομένων, άρα χρειαζόμαστε περισσότερα δεδομένα και χρειαζόμαστε ε, κονδύλια και όχι περικοπές. Όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι, υπάρχει μείωση κατά 44,6% για τον οργανισμό ελέγχου, που είναι ένα από τα πιο σημαντικά μας εργαλεία κατά τη παράνομη αλίας. Και αυτό είναι πραγματικά λυπηρό. Έχω μία ε, σύντομη πρόταση και δεν ξέρω αν θα έχουμε το χρόνο το Σεπτεμβρίο να έχουμε τροπολογίες. Πάντως για το έγγραφο το οποίο τώρα έχουμε ε, στα χέρια μας, ε, νομίζω ότι είναι το σημείο 2 των προτάσεων. Ε, δεν μου αρέσει πολύ η διατύπωση. Έτσι όπως διαβάζω τώρα τη δεύτερη πρόταση, φαίνεται ότι έχουμε χρήματα και πρέπει να τα δώσουμε για τις αλληλευτικές συμφωνίες. Κάπως πρέπει να φροντίσουμε τη διατύπωση γιατί δεν είναι χρήματα που πρέπει ούτω ή άλλω να δαπανίσουμε. Πρέπει να τα δαπανίσουμε εφόσον έχουμε σωστέ και αποδοτικέ συμφωνίε. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Δεν ε, εννοούμε ότι πρέπει να δαπανηθούν αυτά τα χρήματα ούτω ή άλλω ε, για το αποθεματικό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πάω πίσω ένα-δύο βήματα, γιατί ανησυχώ πολύ. Ίσως να υπάρχει κάποια παρεξήγηση όσον αφορά τον προπολογισμό και τα ποσά που προτείνονται σε αυτόν. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είμαστε καθόλου ικανοποιημένοι με αυτά που σε δύο εβδομάδες προτίθεται να υιοθετήσει το Συμβούλιο. Αν επιστρέψουμε στο σχέδιο προπολογισμού μας, είναι καλή αφετηρία πάντα. Και αν δούμε τα διάφορα κεφάλαια, διάφορε κατηγορίε, και αν το κάνουμε αυτό εντάχει προτείνω, θα δούμε ότι σχεδόν όλες οι κατηγορίες, όλα τα κεφάλαια έχουν αύξηση και σε ανάληψη υποχρεώσεων και υποχρεώσεων πληρωμών. Ε, ισχύει για το 11.02 αφορά τις δαπάνες αγοράς όπου οι υποχρεώσεις είναι σταθερές αλλά οι πληρωμές αυξάνονται. Διεθνείς αληφτικές συμφωνίες το ποσό που προτείνεται για την ανάληψη υποχρεώσεων και πληρωμών τα ποσά παραμένουν σταθερά Συγγνώμη, για πληρωμέ μειώθηκαν κατά 5 εκατομμύρια, αλλά η ανάληψη υποχρεώσεων παραμένει σταθερό το ποσό. Βέβαια, υπάρχουν μεγάλα ποσά στο αποθεματικό εκεί. 115 εκατομμύρια ευρώ στο αποθεματικό. Το βάλαμε στο αποθεματικό, σύμφωνα όμω με τι διατάξει τη διαθεσμική συμφωνία που προβλέπει ότι θα πρέπει να μπει αυτό το ποσό στο αποθεματικό αν οι συμφωνίε δεν έχουν τεθεί σε ισχύ την πρώτη η Πρώτου ε, του τρέχοντο έτου εκτέ του προπολογισμού. Τώρα, το κεφάλαιο για στενότερο διάλογο με τον τομέα, εκεί έχουμε ακριβώ τα ίδια από όσον αφορά την ανάλυση υποχρεώσεων και αύξηση πληρωμών εν συγκρίση με τον ε, ισχύοντα προπολογισμό. Και αν προχωρήσουμε και δούμε την Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Αλία, έχουμε αύξηση και στην ανάλυση υποχρεώσεων και στι πληρωμέ. Αν δούμε μετά την υποστήριξη για τη διαχείριση των ληφτικών πόρων, βελτίωση των επιστημονικών συμβουλών, συλλογή στοιχείων βασικά, Εκεί έχουμε μία μείωση 500.000 στην πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συγκρίσει με τον ισχύοντα υπολογισμό στην ανάλυση υποχρεώσεων και μία αύξηση σε πληρωμέ. Και στο κεφάλαιο περί ελέγχου, το τελευταίο, έχουμε μία μείωση, μείωση διότι δεν προτείναμε την ανάλυση υποχρεώσεων για τη μίσθωση του σκάφου. Αν δείτε ότι αυτά που για, τα, για τους ελέγχους των μελών, εκεί έχουμε αύξηση. Αυτό είναι το ιστορικό. Και από αυτή τη βάσεω θα πρέπει να δούμε τι τροπολογίε του Συμβουλίου και ναι, ανησυχούμε λόγω των ε, τροπολογιών του Συμβουλίου και είναι αρκετά σίγουρο ότι αυτά που προτείνει το Συμβούλιο θα υιοθετηθούν. Ε, και να σε επιστήσω την προσοχή σε αυτά που προτείνει το Συμβούλιο σαν αφορά την, ε, ε, τον οργανισμό στο Βίγκο. Προτείνουν μια μείωση 250.000, περίπου 250.000 για το διοικητικό προπολογισμό της υπηρεσίας και προτείνουν και μια μείωση στις πληρωμές 1,29 εκατομμύρια και η μείωση πληρωμών 1,29% για τον οργανισμό. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να το αποδεχτούμε. Αν δούμε τώρα τις άλλες τροπολογίες που προτείνονται, η κυρία Ράιμερ αναφέρθηκε στη μείωση που προτείνεται σε αφορά τη διοικητική υποστήριξη για τη συλλογή ε, δεδομένων, 200.000 ευρώ. 200.000 ευρώ δεν φαίνεται σαν μεγάλο ποσό, όσον αφορά το δικό μας υπολογισμό. 200.000 ευρώ είναι πάρα πολύ σημαντικό ποσό αν δει κανείς αυτή τη, αυτό το κονδύλι. Γιατί έχει 450.000 ευρώ αυτό το κονδύλι. Άρα είναι τεράστια περικοπή. Και είναι ένα κονδύλι που προτάθηκε και πέρσι περικοπή από το Συμβούλιο και τότε ήρθα σε αυτή την επιτροπή σας και εξήγησα ότι εμείς χρησιμοποιούμε αυτό το κονδύλι για να χρηματοδοτούμε τον έλεγχο της εφαρμογής των προγραμμάτων συλλογής στοιχείων από τα κράτη-μέλη. Και αυτά είναι χρήματα που χρησιμοποιούνται πάρα πολύ καλά. Αν παρακολουθείτε η χρήση, η εφαρμογή των προγραμμάτων αποτελεσματικότητα, εντοπίζουμε το ταχύτερο δυνατόν τα προβλήματα, άρα μπορούμε να τα διορθώσουμε και τάχιστα και τα κράτη-μέλη δεν καταλήγουν να πρέπει να επιστρέψουν χρήματα στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βεβαίω μα ανησυχούν άλλε περικοπέ, κυρίω η περικοπή των 40 εκατομμυρίων όσον αφορά τι ανλήψει υποχρεώσεων πληρωμών για το ληφτικό ταμείο και οι περικοπές στην ανάληψη υποχρεώσεων και πληρωμών και για τη συλλογή των δεδομένων και για τις οικονομικές συνεισφορές στα προγράμματα ελέγχου των κρατών μελών. Σε τη συλλογή των στοιχείων έχουμε περικοπή 2 εκατομμυρίων ευρώ Θεωρούμε προφανώ ότι αυτό είναι ασφαλμένο. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν τα αναγκαία στοιχεία για να κάνουμε σωστέ προτάσει και στην περίπτωση των ελεγκτικών προγραμμάτων το, η περικοπή που προτείνεται 1,8 εκατομμύρια στην αλεύση υποχρεώσεων και 3,2 εκατομμύρια σε πληρωμέ. Και αυτά δεν μπορούμε να τα υποστηρίξουμε σαν μέτρα. Για να, να πω κάτι για τα πιλωτικά προγράμματα. Υπάρχει ένα πιλωτικό πρόγραμμα που ανέφερε η κυρία Λόουεν το πρόγραμμα για τη μίσθωση σκάφους για επιστημονικούς ελέγχους, επιστημονικές ερεύνες. Είμαστε πεπισμένοι ότι χρειάζεται να ενισχυθεί, να αυξηθεί η επιστημονική μας γνώση όσον αφορά τις αληφτικές συμφωνίες που συνάπτουμε. Θέλουμε να αλλιεύουμε μόνο από το πλεόνασμα και χρειάζεται να έχουμε τις σωστές επιστημονικές πληροφορίες γι' αυτό. Δεν είμαστε σίγουροι κατά πόσο η μίσθωση ενός σκάφους είναι η σωστή προσέγγιση. Δεν είμαστε σίγουροι ότι έτσι θα επιτεθούμε μακροπρόθεσμα κατά του διαθωτικού προβλήματος. Θέλουμε να υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας με κάποιους περιφερειακούς οργανισμούς της Δυτικής Αφρικής, κάτι που ήδη μπορούμε να τα κάνουμε σύμφωνα με το δεύτερο μέσο που διαθέτουμε, αλλά ίσως να μην έχουμε αρκετούς ε, πόρους για να το κάνουμε αυτό. Θέλουμε να επιστρέψουμε, να το συζητήσουμε ξανά με την κυρία Λόβεν αυτό το θέμα, αυτή την πρόταση, για να μπούμε σε περισσότερες ε, λεπτομέρειες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Yeah. Äh, σας ευχαριστώ πολύ για τις παρεμβάσεις σας. Ήταν ενδιαφέρον να ακούσω τις απόψεις σας. Νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό συμφωνούμε. Δεν θέλουμε να έχουμε μείωση των δαπανών για τον έλεγχο. Η πρόταση της κυρίας Λεωβίνη είναι πολύ ενδιαφέρουσα και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το συζητήσουμε πολύ προσεκτικά, να δούμε πώς θα βρούμε τους κατάλληλους πόρους. Γιατί είναι δύσκολο να πείσουμε το Συμβούλιο να απελευθερώσει πόρους συμφωνούμε, όπως σας είπα, ότι δεν πρέπει να μειώσουμε ε, τα κονδύλια για τον οργανισμό, γιατί εκεί πρέπει να επιτύχουμε και κάποια πρόοδο στο να περιορίσουμε την παράνομη αλία, όπου συνεχίζουμε να έχουμε μεγάλα προβλήματα. Και εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ περιοριστικό το Συμβούλιο και γι' αυτό θα πρέπει να προσέξουμε να μην επηρεάσουμε μελλοντικέ ε, πολιτικές, ε, μελλοντικά προγράμματα στον τομέα της αλίας Πρέπει να επιτρέψουμε να υπάρχουν οι κατάλληλοι πόροι και για μελλοντικέ ε, πολιτικές και γι' αυτό θέλουμε να παραμείνει και ε, η χρηματοδότηση του οργανισμού. για τις υφιστάμενες συμφωνίες ε, θα πρέπει να συνεχίσουμε να διαθέτουμε τους κατάλληλους πόρους. Δεν μπορούμε να υπαναχωρήσουμε επί συμφωνιών που ήδη έχουμε συνάψει. Πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι αυτοί. Και αυτό που αναφέρουμε για το αποθεματικό δεν σημαίνει ότι πρέπει να δαπανηθούν τα χρήματα. Θα πρέπει να βρούμε την κατάλληλη διατύπωση, γιατί νομίζω θα συμφωνήσουμε σε αυτό το σημείο. Απλώ είναι θέμα διατύπωση. Ευχαριστώ. Κύριε Ρέιμερς, μια ερώτηση. Εδώ έχω τη θέση σας ως εισηγήτρια και δεν είστε κατά όλων των στοιχείων που έχει το σχέδιο του προπολογισμού. Σωστά τα λέω. Τα στοιχεία λοιπόν που έχω εδώ δεν συμπίπτουν με το προσχέδιο του προπολογισμού που έχει η Κομισιόν. Εσείς θα αντιταχθείτε σε όλα αυτά τα στοιχεία που αναφέρει το προσχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υποστηρίζω την Επιτροπή. Νομίζω ότι το είπα αυτό. Με το Συμβούλιο έχουμε μεγαλύτερες διαφορές. Στα συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία, αυτό που έκανα ε, είναι να δώσω τα, τα στοιχεία και νομίζω ότι το βλέπετε. Είναι διαθέσιμα αυτά τα στοιχεία, μπορείτε να τα δείτε τα αριθμητικά δεδομένα. Eh. Ναι. Στα διοικητικά θέματα εσείς συμφωνείτε με το Συμβουλίο. Πάντως, ε, όπως ρώτησα, δεν είστε κατά των στοιχείων που αναφέρει η Κομισιόν, έτσι δεν είναι. Εγώ ήθελα να το διευκρινίσω αυτό γιατί δεν το είχα καταλάβει. Ε, Εκεί που συμφωνεί το Συμβούλιο με την Επιτροπή, υποστηρίζουμε το Συμβούλιο, την Επιτροπή, συγγνώμη, αλλά υποστηρίζουμε και το Συμβούλιο. Εκεί που υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ Συμβουλίου και προτάσεων της Επιτροπής, εκεί διαφοροποιούμε από τη θέση του Συμβουλίου. Δεν καταλαβαίνω το πρόβλημα. Υποστηρίζω την Επιτροπή. Αν και το Συμβούλιο έχει την ίδια θέση με την Επιτροπή, τότε υποστηρίζω και το Συμβούλιο. Εκτό από τα σημεία στα οποία διήσατε οι απόψει του, όπως σας είπα. Συγγνώμη, ε. δεν θέλω να είμαι σχολαστική, αλλά σε κάποια σημεία υποστηρίζετε την Κομισιόν, αλλά για τις δικέ δαπάνες, τις πρώτες ε, δημοσιονομικέ γραμμέ, δεν την υποστηρίζετε. Αυτό το, γι' αυτό επιμένω. Τα αρχικά στοιχεία, το ξαναλέω, δεν συμπίπτουν. Αλλά εντάξει, δεν θα επιμένω για να μην κάνουμε τώρα μεγάλη σύστηση για αυτό το θέμα. Πάντως, ολοκληρώσαμε και με το σημείο αυτό της ημερήσιας διάταξης, το 7. Έτσι δεν είναι. Τελειώσαμε λοιπόν με αυτό το σημείο 7 της ημερήσιας. Τροπολογία για η ημερομηνία, συγγνώμη, για τις τροπολογίες είναι 20 Ιουλίου, 12 το μεσημέρι. Αλλά γι' αυτό ρώτησα για τα στοιχεία προηγουμένω στην εισηγήτρια, για να δούμε κατά πόσο είμαστε αντίθετοι σε όλα τα στοιχεία τη Κομισιόν. Διαφορετικά θα πρέπει να πάμε σε προφορικέ τροπολογίε τη ημέρα τη ψηφοφορία, το οποίο θα είναι χαόδε. Τέλο πάντων, 20 Ιουλίου, την προμηνία κατάθεση των τροπολογιών, 12 το μεσημέρι. Αλλά έτσι φαίνεται να λειτουργεί. Χαοτικά δηλαδή ο προπολογισμό φέτο για όλα τα θέματα με τροπολογίε τελευταία στιγμή και δεν μπορούμε να προχωράμε έτσι. Εντάξει, δεν θέλω να κάνω την γκρινιάρα, είμαι και παλιά στο κοινοβούλιο, αλλά αυτά δεν τα καλοβλέπω. Τελειώσαμε τέλο πάντων το σημείο 7 τη ημερήσια και περνάμε στην ανταλλαγή απόψεων με εκπρόσωπο τη Επιτροπή σχετικά με τις συμφωνίες αλληλείας με τρίτες χώρες και τις διαπραγματεύσεις ανεξελίξη και κλεισμένων των θυρών. Παρακαλώ όσοι δεν είναι βουλευτές να εξέλθουν και ο εκπρόσωπος Κομισιόν να έρθει εδώ.